πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα. Η Γκουε μου ζήτησε τον διορισμό μελών σε κάποιες από τις αντιπροσωπείες και από τις ε, επιτροπές. Βεβαίως αυτό θα εγγραφεί στα πράγματα.